Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε με τις προφορίες. Το πρώτο μας σημείο, πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, που τροποποιεί την οδηγία για τα απόβλητα. Η κυρία Σιμώνα Μποναφέ, εισηγήτρια. Λοιπόν, το πρώτο είναι η 366, τροπολογία 366 υπέρ, 366 υπέρ, κατά, για να ελέγξουμε. 366. Πρόεδρε, μια ερώτηση. Ποια Ποια τροπολογία ψηφίζουμε. Την πρώτη. 366. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα είναι... Υπέρ. Εγκρίνεται. 367. Ωραία, ξαναψηφίσουμε 366, αφού λέτε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι, κυρία Στίβενς. Με συγχωρείτε. Ο συνάδελφος δεν είναι εδώ, ε, μάλλον η κάρτα μου δεν είναι εδώ, την έχει πάρει ένα συνάδελφος για άλλη επιτροπή. Θα μου τη φέρουν. Mijn stemkaart is onderweg. Έρχεται, έρχεται, θα ψηφίσω εντός ολίγου. Then you πείτε τι ψηφίζετε και θα σας ε, λάβουμε υπόψη. Να ξαναψηφίσουμε την 366. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κυρία Στίβενς είναι υπέρ. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 367 υπέρ κατά Συμβιβαστική συμβαστική 1α υπέρ κατά απορρίπτεται νομίζω αλλά σε ελέγξουμε διότι είναι συμβαστική Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1B. Η 1B καταπίπτει. Συμβαστική 50. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 370 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ήτρε 33 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Θα πρέπει να συνηθίσω τα χρώματα. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 423. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 436. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 39. Υπέρ. Να ελέγξουμε. 436. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω σχεδόν όλοι κατάψηφισαν, αλλά τέλο πάντων. Όπω βλέπετε κι εσεί, απορρίφθηκε. Ήτρε 39. Ήτρε 39 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ήτρε 40 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 43 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 492 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 493. Καταπεπτεί. Ωραία, να πάμε στη συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 46. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57. Καταπίπτει. Καταπίπτει, καταπίπτει. 510 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 511 πανομοιότυπη. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 514 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 516 και 517 από κοινού. Υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 5-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Θέλετε να, ψη... να ελέγξουμε για την 5-18. Άντε, ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. 58 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 519. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την 532. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, την ψηφίζουμε μαζί με την προφορική. 5.32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 607 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 609 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 608 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 646 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, Κάτι μα ξέφυγε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πολύ κύριε Ντέμεσμακερ. 6.59. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 731 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 827. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ήταν πολύ καλή συμβαστική συνάδελφοι. Σελίδα 69. 460 υπέρ. Κατά αποχές εγκρι... Ε, απορρίπτεται. 459 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 47. Α, ήταν πανομοιότυπη μάλλον. 515 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 457 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εντάξει, 457 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Καλά που μου το είπατε. 959 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Έλεγχο. Ας ελέγξουμε. Ελεκτρονική ψηφοφορία 959. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρέπει να δω καλύτερα τις πλειοψηφίες εδώ πέρα. Συμβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 καταπίπτουν. Συμβαστική 31 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 994 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35, συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1009 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10-12, 1012. Θέλετε να Ελέγξουμε τη 1009. Ψηφίζουμε για το 1009. Πέρας. Και εγκρίνεται. 1012. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καλά να ελέγξουμε. Πέρας, απορρίπτεται. Συμβαστική 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 74 υπέρ, κατά αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ, έλεγχο, έλεγχο για την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Συμβαστική 47 υπέρ. Παρακαλώ να σκόλετε τα χέρια σας. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 1054 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1056 και 57 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 92 την ψηφίσουμε, κατέπεσε. κατέπεσε. Συμβαστική 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 44. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1171-1171 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος. Πέρας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εγκρίνεται. 1173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 1176 υπέρ. Ξανά υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 1177 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1178 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε αν θέλετε. 1180. 1180. Πέρας. Απορρίφθηκε. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 1182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1183 υπέρ. Α, κατέπεσε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «1142 και 102 ε, μαζί, υπερκατάποχες εγκρίνονται, 1235 ε, και 1236 μαζί, υπέρ. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ήταν σχετικά σαφές αυτή τη φορά, αλλά σε ελέγξουμε. και 1236, πέρασε. Εγκρίθηκε. 1239 και 1240 και 1241 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 1242 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1243 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1243, 143 μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1244 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 1246 και 1247 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ήτρε 103. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1249. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1250. ...1250 υπέρ, κατά, Νομίζω ότι απορρίφθηκε, να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτω. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 51. Υπέρ. Κατά. κατά, Αγκρίνεται. Τροπολογία 1258. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Συμβαστική 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Συμβαστική 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 1284. 1284. 1284 υπέρ. Κατά. Αποχές. ογδόντα 1286 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1294. 1294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1300 και 1301 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1302. Την ψηφίσουμε. Ωραία. 1302. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 75, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 58, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 193, υπέρ, α, Επίδειξα μια συμβαστική. Συμβαστική 78. 78 υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 193 υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 59 υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Έχουμε μια σειρά από πανομοιότυπε τροπολογίε. 198, ή 6, 204, 228, 227 και. και οι άλλοι όχι. Ψηφίζουμε όλε αυτέ Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 215. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμμεβαστική 60. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 61 Συμβαστική 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 226. Πέρας. Εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 252. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 253 υπέρ. Υπέρ της 253. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 76. Θέλετε έλεγχο. Ήταν κοντά τα αποτελέσματα, αλλά ας ελέγξουμε. Εγώ νομίζω ότι εγκρίθηκε. 253. Πέρας. Ναι, εγκρίνεται. Συμβαστική 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. 265. Πέρας. Εγκρίνεται. 266 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύπτεται. 267. Υπέρ. Κατά. 267. Τα πολύ γρήγορα. 273. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 276 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 καταπληκτή Α, την ψηφίζουμε. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 279 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 282 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 283 κατά καταπιπτή. 287, 287 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές. Δεν είμαι βέβαια γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Να ψηφίσουμε. Για την Ήτρε 17. Πέρας. Ήταν πολύ κοντά τα αποτελέσματα. Απορρίφθηκε. να μια ψήφο διαφορά. Συμβαστική 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 24 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 327 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70, συμβαστική 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 351 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 352 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 358 υπέρ. Ξανά. 358 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. ξεκάθαρα εγκρίνεται. Συμβαστική 72. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 73. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 364. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ήτρε 30. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ήτρε 31. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεν ψηφίζετε. Δίκη σας επιλογή. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι στην εισηγήτρια. Και σε όλους όσοι εργάστηκαν για το σημαντικό αυτό θέμα. Επόμενο. Έρχεται, έρχεται. we start Αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενη ψηφοφορία για τους χώρους ταφής υγειονομικών, ε, χώρους υγειονομικής ταφής Παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε ένα λεπτό, λέει ο κύριος Λίζε, για να διανύμουμε τον επόμενο κατάλογο ψηφοφορία, γιατί πήγατε πολύ γρήγορα. Ναι, κάντε με ένα νόημα, λέει πρόεδρος. Είναι λοιπόν το επόμενο θέμα. Οι χωματερές, προετοιμαστείτε. Είμαστε εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Κύριε Μποναφέ, είναι η συγγήτρια. Πρόταση οδηγίας Ξεκινήσουμε, ξεκινάμε τροπολογία 85 υπέρ. 85 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε όμως. Okay. On 85. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 89 απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πού πάμε τώρα 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Όχι συζητώ, συγγνώμη. Τροπολογία 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ όχι καταπίπτει. Δεν καταπίπτει. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 λέει, πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ή 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163-164 ταυτόσμες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πηγαίνουμε σε τολικές αναφορές 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Και η τρένα. Κατά πίπτου. 35. Και αυτή. Και 36. Ψηφίζουμε την 37. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ψήφι Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα. Έλξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Καλά κάνουμε και ελέγξαμε. Ήτρε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τοπλογία 50 κατά πίπτη που πηγαίνουμε στην Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά Αποχές. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Γιατί κάποιοι δεν σηκώσουν τα χέρια. 72. Έλεγχος. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήτρε 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Ήτρε 10. πέρες ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψήφι υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται. Ήτρε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της δύο εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος τώρα. Α, εδώ έχουμε μια τροπολογία. Την υπαριθμό 30. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι στην κυρία Μοναφέ και σε όλους τους υπολείπους που εργάστηκαν για αυτό το έγγραφο. Επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο οδηγίας για το WIT Μποναφέ και πάλι. Η συγγήτρια 39 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 1 υπέρ. και 1. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 και ήτρε 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται ήτρα 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρα 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 και η 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 72 και η 34. υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 73 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ή 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 και η 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 27 υπέρ Ήτρε 27. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 80 και 29 υπέρ κατά ποχές απορρίπτονται 81 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 96 και 98 υπέρ κατά εποχές απορρίπτονται 97 και 99 υπέρ κατά εποχές απορρίπτονται 20 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται οι 3 2 ήταν μαζί ναι 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ήτρε 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 30 κατά 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καλώς και πάλι 31. Υπέρ. Αρχίστε να σηκώσετε τα χέρια σας, αυτό εγώ. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, ευχαριστώ. Ήτρε 5, καταπίπτει. Ήτρε 6, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 ή 37 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τι δύο την ψηφίζουμε, ναι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, όχι, καταπίπτει. Επειδή εγκρίθηκε 2, έτσι μάλιστα. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και Τέλος, το σύνολο του σχεδίου έκθεση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Τώρα ψηφίζουμε κάποιες τροπολογίες. Ναι, ορίστε. Ναι. Στο σχέδιο θετικού ψηφίσματος. Ή τρένα. Πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Όχι. Ήταν ταυτόσιμη, συγγνώμη. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήστε και Μποναφέ. Και όλους τους υπολείπους που εργάστηκαν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ in the afternoon is We could have done something more. It's just yes. you went so fast. they uh, so, dear colleagues, uh... Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Για σήμερα το πρωί θα επανέλθουμε το απόγευμα. Εάν είχατε το κατάλογο των ε, ψηφοφοριών ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Διακόπτουμε μέχρι τις 11 όπου θα έχουμε τον Υπουργό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μάλτας. Σας ευχαριστώ.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

Hello, Αγαπητοί συνάδελφοι. Uh, Προτείνω να συνεχίσουμε. Καλώ uh, to welcome. ορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Μαλτέζικης Προεδρίας, τον Υπουργό κ. Χερέρα, που βρίσκεται εδώ σήμερα για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ε, θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much. First of all, I take the Σας ευχαριστώ κυρία Βαλεάν. Καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ε, στη θέση της Προέδρου της ε, Εξαιρετικής Αυτής Επιτροπής. Θα μιλήσω λίγο μαλτέζικα και μετά θα επανέλθω στα αγγλικά. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας και να συζητήσω μαζί σας πιο αναλυτικά τη δουλειά που μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Όπως θα δείτε, η Μαλτέζικη Προεδρία θα προσπαθήσει να τοποθετήσει πάλι τον πολίτη στο επίκεντρο της Ευρώπης. Η Επιτροπή σας ασχολείται με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ε, το περιβάλλον, ε, την ασφάλεια τροφίμων. Είναι όλα θέματα που επηρεάζουν άμεσα την ευημερία των πολιτών και έχουμε να παίξουμε ζωτικό ρόλο εάν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Τα τελευταία 60 χρόνια η Ευρώπη θεωρήθηκε υπόδειγμα ελπίδας, ευημερίας, ανάπτυξης και ειρήνης. Αυτό ήταν ε, ε, κατόρθωμα των πρωτοπόρων του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ε, σε εποχές που υπήρχε σκεπτικισμό σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό μαζί. Τώρα, στην 60η επέτειο του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματο, Μάλτα έχει την τιμή να προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργών και θα πρέπει να κοιτάξουμε τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τα όσα έχουμε πετύχει και να μεταφέρουμε τα πλεονεκτήματα αυτού του κατορθώματος στους πολίτες μας. Πλεονεκτήματα τα οποία συχνά ξεχνιόνται. Επίσης είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε το μέλλον. Η Ευρώπη χρειάζεται νέα ορμή. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν δείξει σαφώς την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και να μεταφέρει πιο αποτελεσματικά να μεταδώσει τα μέτρα που λαμβάνει για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της. Τα πολιτικά γεγονότα της περσινής χρονιάς έχουν σημαδέψει όλους μας. Ποτέ στο παρελθόν δεν χρειαζόμασταν μεταρρύθμιση τόσο πολύ όσο τώρα, ούτε χρειαζόταν να είμαστε τόσο κοντά στους πολίτες μας όσο τώρα. Πέρσι σύστηκαν τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Εχειρήματο. Η Μάλτα είναι αποφασισμένη να συμβάλλει στην επιτυχία της Ευρώπης. Θα καταβάλουμε προσπάθειες στο Συμβούλιο και σε συνεργασία μαζί σας Ελπίζουμε να έχουμε πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι μήνες είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε φιλόδοξους στόχους. Και για να προωθήσουμε ε, τις φιλοδοξίες μας ε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει επίσης ε, να γνωρίζουμε πού στοχεύουμε. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς διαμεσολαβητές ε, χωρίς ε, κρυμμένο θεματολόγιο. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πνεύμα συνεργασίας ε, και ειλικρίνειας. Ο Πρωθυπουργός, ο αναπληρωτής πρωθυπουργό, ο υπουργό οικονομικών, όλοι υπήρξαν ευρωβουλευτέ και γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι ε, να νομοθετούμε προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Με την συνθήκη της Λισαβόνας, ε, το Κοινοβούλιο έχει εξίσου πολύ εξουσία με το Συμβούλιο. Προσλέπω στην καλή συνεργασία μαζί σας πάνω στα πιο σημαντικά θέματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι μεγάλη μας τιμή να προεδρεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη κρίσιμη χρονική στιγμή. Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές μας ε, θα είναι η προσπάθεια να δώσουμε περισσότερη ορμή στις εργασίες και να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσουμε το βιωτικό τους επίπεδο. Έχουμε εντοπίσει έξι προτεραιότητες, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την ενιαία αγορά, την πολιτική γειτονία, σε την κοινωνική ένταξη ε, και ναυτιλιακά. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο, εάν μου επιτρέπετε, κυρία Βάλιαν, θα ήθελα να μιλήσω ε, για τα θέματα που αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής σας. Κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ τώρα λοιπόν στις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας που σχετίζονται με τις εργασίες της Επιτροπής σας. Καταρχάς όμως να ε, σας πω πώς θα προχωρήσουμε. Εγώ θα καλύψω το περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος, φυτοϊγειονομικά θέματα, ενώ ο συνάδελφός μου Κρίς Φέρν θα ασχοληθεί με την δημόσια υγεία και το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας. Είναι πρώτη φορά που η Μάλτα κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή, αποτελεί και πρόκληση. Έχουμε κάνει εκτενείς προετοιμασίες και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ισχυρό θεματολόγιο το οποίο θα μπορέσει να βελτιώσει τις πολιτικές ε, περιβάλλοντος, αντιμετώπιση αλλαγής του κλίματος ε, και φυτογενομικών θεμάτων. Ε, συνεργαζόμαστε στενά και με τους εταίρους μας στο τρίο προεδριών της κατοχώρες και την Σλοβακία και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την καλή συνεργασία μαζί τους. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια από τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας αλλαγή του κλίματος, ε, κυκλική οικονομία, ε, θεματολόγιο 2030 ε, και μικροβιακή αντοχή. Καταρχάς λοιπόν όσον αφορά την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Με την Συμφωνία του Παρισιού, που έχει τεθεί σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ε, στην κορυφή της ε, διεθνούς ε, διαδικασίας. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι έφραυστη και θα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρηθεί η ορμή που έχει δοθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ηγείται δίνοντας το καλό παράδειγμα και να είναι φιλόδοξος και αξιόπιστος διαπραγματευτής, συνομιλητής στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δίνουμε προτεραιότητα στο σύστημα ε, πορείας εκπομπών ε, καθώς ε, και σε θέματα εκτός από αυτό. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος μέχρι το 2030. Καταλαβαίνουμε ότι ένα στεναρό σύστημα που να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις ε, ε, για χαμηλές εκπομπές ε, άνθρακα είναι απαραίτητο. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να απλοποιηθεί χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Ως Προεδρία Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, οι οποίες ε, θα βασίζονται στην πρόοδο που σημειώθηκε επί Σλοβακικής Προεδρίας ε, για να πετύχουμε κοινή προσέγγιση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κύριο Ντάνκαν για την επιτυχή ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή. Η Μαλτέζικη Προεδρία επίσης ε, θα προσπαθήσει να πετύχει πρόοδο πάνω στον ε, κανονισμό για τον ε, επιμερισμό της προσπάθειας για τη μείωση των εκπομπών. Και εδώ πάλι ο στόχος μας θα είναι να βασιστούμε στην καλή δουλειά που έκανε η Σλοβακική Προεδρία. Επίσης, ε, οι εργασίες ε, πάνω στην πρόταση αυτή θα ε, συμπληρωθούν από προσπάθειες πάνω στην πρόταση Λούλου για την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να πετύχουμε τις φιλοδοξίες μας όσον αφορά την, το μετριασμό της αλλαγής ε, του κλίματος. Οι συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε θέματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναλύουμε ε, μέσα στους επόμενους μήνες για να πετύχουμε κοινή θέση πάνω στην πρόταση της ε, Κομισιόν ε, στο Συμβούλιο ε, της 19ης Ιουνίου του 2017. Επίσης, η Προεδρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλο ενδιαφέρον και προσλέπουμε σε περαιτέρω επαφές στο μέλλον. Άλλο σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τα αποτελέσματα της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης ΙΚΑΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την συμπερίληψη ε, της ε, αεροπλοείας ε, στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Προσλέπουμε λοιπόν στην πρόταση αυτή και είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε επικοδομητικά με το Κοινοβούλιο με βάση την δεύτερη αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η κυκλική οικονομία. Πρέπει να ε, τονίσουμε την ε, δέσμευση του Συμβουλίου για μετάβαση σε κυκλική οικονομία όσο γίνεται πιο γρήγορα με βάση τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν ε, τον Ιούνιο του 2016. Τα πιθανά πλεονεκτήματα τη κυκλική οικονομία είναι τεράστια και πιστεύουμε ότι το πακέτο, η δέσμη μέτρων τη Κομισιόν θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προ ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο πρότυπο. Επίσης, ε, η καλή διαχείριση αποβλήτων ε, είναι απαραίτητη για να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Η Μαλτέζικη Προεδρία θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στο θέμα αυτό εντός του Συμβουλίου. Σκοπεύουμε να βασιστούμε στην ε, σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Προεδριών. Επίσης, η Προεδρία είναι διατεθειμένη να συνεχίσει εξίσου εντατικά τις εργασίες και να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, κατά την πρώτη ανάγνωση. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μποναφέ που κάθεται εδώ μπροστά. διότι έμαθα ότι η ψηφοφορία σήμερα διεξήχθη πολύ καλά. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνάντηση κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών ε, του Σεπτεμβρίου του 2015 είναι γεγονό το οποίο θα πρέπει να δοθεί συνέχεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030. Καταλαβαίνουμε ότι απομένει αρκετή δουλειά να γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε πολλούς τομείς πολιτικής. Γι' αυτό στις 19 ε, Σεπτεμβρίου είχαμε την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο «Δεπόμενα βήματα για τη βιώσιμη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή δράση για βιωσιμότητα». Ε, η οποία παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Η Μαλτέζικη Προεδρία ε, έχει προγραμματίσει υπουργική συζήτηση κατά το επόμενο Συμβούλιο Περιβάλλοντος ε, τον Φεβρουάριο, που στόχο έχει να επικεντρωθεί και στην εφαρμογή του θεματολογίου 2030 και συγκεκριμένα ε, στην ε, πολιτική περιβάλλοντος. Η Προεδρία επίσης στόχο έχει να υιοθετήσει συμπεράσματα τον Ιούνιο κατά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, για να δώσει μια συνολική απάντηση στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, γνωρίζουμε ότι η Προεδρία μας πραγματοποιείται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την μικροβιακή ε, αντοχή και την απειλή της, ε, ε, στην υγεία των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αναθεωρημένο σχέδιο δράσης ε, για τη μικροβιακή αντοχή, μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας, που θα βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μικροβιακή αντοχή, που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2016. Θα διασφαλίσουμε έτσι το Συμβούλιο να συνεχίσει να είναι ενεργός παραγοντα στο θέμα αυτό. Επίσης ε, σημαντικά θέματα είναι οι φαρμακούχες ζωοτροφές εδώ. Ε, έτσι μπορούμε να πετύχουμε συγκεκριμένη και απτή πρόοδο στα θέματα αυτά. Κυρίες και κύριοι, πέρα από τα θέματα που ήδη ανέφερα, θα δώσουμε σημασία και σε κάποια άλλα θέματα που παραμένουν επιτάπητος. Ε, θα ολοκληρώσουμε ε, την ε, συμφωνία του ε, Γκέτεμπορκ, καθώς ε, και το θέμα του υδραργύρου. Θα ήθελα να αναγνωρίσω τις επιτυχείς προσπάθειες της Σλοβακικής Προεδρίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή Στέφαν Εκ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, πρώτη ανάγνωση πάνω στο θέμα αυτό και θα ε, εργαστούμε με στόχο την υιοθέτηση ε, του θέματος αυτού εγκαίρως για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πραγματοποιηθεί στην πρώτη διάσκεψη των μερών το καλοκαίρι. Άλλο θέμα που έχουμε ακόμα είναι η αναθεώρηση του κανονισμού για το Euro 56. Και επίσης έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την ε, αξιολόγηση της εφαρμογής τους. 28 Φεβρουαρίου έχουμε συζήτηση των Υπουργών ε, για να συμβάλλουμε στο πρασίνισμα του ευρωπαϊκού εξαμείνουν την περιβαλλοντική κατεύθυνση δηλαδή. Και επίσης το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2015 υπογράμμισε την ε, σημασία να διατηρηθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και να μην ε, μειωθεί ε, το επίπεδο. Και ακριβώς γι' αυτό επικροτώ τα αποτελέσματα του REFIT. Ωστόσο, Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, απομένει να γίνει πολλή δουλειά, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή και καλύτερη συνεκτικότητα ανάμεσα στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Συμβούλιο και η Προεδρία προσβλέπουμε λοιπόν ε, στο επόμενο σχέδιο δράσης. Τέλος, ε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Υπουργική Συνάντηση 25 και 26 Απριλίου στην Βαλέτα, όπου θα επικεντρωθούμε στο κλίμα, ε, θέματα ε, ναυτιλιακά, τα πλαστικά και την ε, και τον τρόπο που επηρεάζουν οι πολιτικές μας το θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν το θεματολόγιο για την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και προσβλέπω σε επικοδομητικές συζητήσεις πάνω στα σημαντικά αυτά θέματα να σημειωθεί ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ε, σε συνέχεια συνάντησης ε, για αναστηλιακά θέματα στην ε, Μάλτα, στο όπου ελπίζουμε να πετύχουμε πλεονεκτήματα και για άλλους τομείς πέρα από τον τομέα των ε, υδάτων. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε εκπονήσει ένα εκτενές θεματολόγιο για την Προεδρία μας. Ε, προσλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για να πετύχουμε αυτή πρόοδο ε, σε μια σειρά πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, υγεία, ασφάλεια και το βιωτικό επίπεδο των ε, Ευρωπαίων πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Πολύ άρτια και φιλόδοξη η ατζέντα, το θεματολόγιο σας και ελπίζουμε πραγματικά να έχουμε νομοθεσία για το καλό των πολιτών και των χωρών μας τώρα να παρακάσω τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Ξεκινώ σύντομα με τους συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο, να κάνει ερωτήσεις, σχόλια. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε συμφωνήσει ως προς το χρόνο δύο λεπτά αρχικά για κάθε μιλητή με πρώτον εκ μέρους του ΕΛΚΑ τον κύριο Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Ερέρα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Συγχαρητήρια για την Προεδρία και ε, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην χώρα σας προς ε, το συμφέρον βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για τη Συμφωνία των Παρισίων που αναφερθήκατε είναι τα πράγματα ε, πολύ λεπτά και δεν μιλώ μόνο για τη ΣΥΠΑ, αλλά έχουμε το κλίμα, έχουμε την ενέργεια, ε, την εξάρτηση από την λοιπά. Το ETS ε, είπατε ότι είναι ένα από τα βασικά συστήματα που θα σας απασχολήσουν. Όπως γνωρίζετε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω τουλάχιστον ότι θέτησαμε μια καλή συμβαστική πρόταση στην Επιτροπή μας, η οποία θα συζητηθεί στο, στο Ολομέλη του Φεβρουαρίου θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια από πλευρά σα. Ποια είναι η άποψή σα για αυτό που εγκρίναμε εδώ εμεί στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή έχουμε φιλοδοξία για να μειώσουμε του, τις εκπομπές MSA αλλά και να προστατεύσουμε από την διαρροή άνθρακα. Και ειδικά σε ό,τι αφορά αυτό το μοντέλο διαρροής άνθρακα που εγκρίθηκε στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς ε, τι άποψη έχετε ως προς το κείμενο αυτό, η φιλοδοξία είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά MSR και η αντιστάθμιση των έμεσων ταπανών έμεσου κόστους, κάτι πολύ σημαντικό για πολλούς. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ισορροπημένοι στις αποφάσεις μας, υπάρχουν επίσης επιτάπτως κάποιες προτάσεις αλλά και αποφάσεις σε ό,τι αφορά τομεακά ή διατομεακά τη μείωση και την προσαρμογή των εκπομπών. Αεροπορία. Μιλήσε το μηχανισμό Stop the Clock που πλησιάζει. Περιμένουμε και την πρόταση της Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη, σύντομα δηλαδή. Θα είστε ένας έμπιστος ε, συνομιλητής και διαμεσολαβητής. Η πρόταση έχει κατατεθεί τουλάχιστον 5% των ευρωπαϊκών πτήσεων να ενταχθούν στην πρόταση ETS. Είναι καλή αυτή η εξέλιξη κατά την άποψή σα και είναι έτοιμο το Συμβούλιο να το υποστηρίξει αυτό. Και κάτι αντίστοιχο, και είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, σε ό,τι αφορά την αυσιπλοεία σαφής η θέση της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Θέλουμε να τονωθεί ο τομέας, να μειωθούν εκπομπές, να υπάρξει ένα είδος αυτορύθμισης στο πλαίσιο του κλάδου. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, στις αρχές της επόμενης δεκαετίας η Ευρωπαϊκή αναυσιπλοεία θα πρέπει να ενταχθεί στο CTS αν συμφωνείτε βέβαια, ποια είναι η δική σας άποψη για όλες αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ κύριε Αντάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Υπουργό Χερέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Από πλευράς μου μελέτησα τις προτεραιότητες όπως υποβλήθηκαν από την Μαλτέζικη Προεδρία στο χώρο που μας ενδιαφέρει και από τον ίδιο τον Υπουργό και αυτό που χρειαζόμαστε είναι χειροπιαστά αποτελέσματα για να προχωρήσει η Ευρώπη προς την ε, διεύρυνση που θα έχει επικεντρωθεί στην ε, συμμετοχή των πολιτών, την καλή τους υγεία και την βιωσιμότητα. Ήθελα να αναφερθώ και εγώ στη Συμφωνία των Παρισίων, όπως και ο συνάδελφος, διότι πιστεύω ότι αυτή η Προεδρία μπορεί να συνεχίσει να αξιοποιεί τον απόϊχο που έχει αφήσει η έγκριση της ε, Συμφωνία των Παρισίων και μετά τη Σύνοδο του Μαρακές ελπίζουμε ότι με τη Συμφωνία UNFCC θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα για τις κλιματικές αλλαγές και το θέμα της ενέργειας. Εδώ λοιπόν έρχονται και ερωτήσεις που ε, θέλω να σας θέσω Υπουργέ να ταιριάξουν. Δηλαδή για το κλίμα. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Μαλτέζικης Προεδρίας σε σχέση με την προσαρμογή και τη στρατηγική της. Και σε σχέση με αυτό, σε ό,τι αφορά την ε, νομοθεσία, νομοθεσία που είναι πολύ σημαντική για μα ε, στο Κοινοβούλιο και έχουν να κάνουν με τις κλιματικές αλλαγές. Το σύστημα ανταλλαγής εμπορία εκπομπών, δικαιωμάτων ε, εμπορία εκπομπών, έχει να κάνει και με τον επιμερισμό τη ευθύνη του βάρους. Πώς θα προχωρήσουν τα δύο αυτά νομοθετήματα παράλληλα, τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία. Και Πώ βλέπετε το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ε, τριών θεσμικών οργάνων. Επίσης θέλω να αναφερθώ και σε κάτι που και εσείς θίξατε. Η Μαλτέζικη Προεδρία λέει ότι θέλει να διερευνήσει τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας για το Euro 5 και Euro 6, ένα ντοσιέ που μα απασχολεί εδώ και καιρό και αυτό το βρίσκω πολύ θετικό. Θέλουμε να κλείσει αυτό το θέμα, το θέμα μείωση των εκπομπών των αυτοκινήτων και πραγματικά θέλουμε να ξέρουμε ποιε είναι οι συγκεκριμένε ε, φιλοδοξίε τη ε, Προεδρία σχετικά για να έχουμε και τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Η κυρία Γκέρλινγκ. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε Υπουργέ Ήθελα να θέσω ερωτήσεις για δύο θέματα. Πρώτον, και όλος ιδιαίτερος να ευχαριστήσω εσάς και τον Πρωθυπουργό σας για την ομιλία του της Ολομέλειας την προηγούμενη εβδομάδα όταν αναφέρθηκε στο Brexit και τόνισε πως ο στενούς ιστορικούς δεσμούς έχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μάλτα. Ήταν πολύ μετροπαθή στι δηλώσεις του και ελπίζω έτσι να ήταν και όσοι τοποθετούνται για το θέμα αυτό. Επ' αυτού λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε στο επίπεδο του Συμβουλίου. Θα γνωρίζετε ότι εμείς εδώ στην Επιτροπή μας και σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο Βλέπουμε ήδη τι επιπτώσει του Brexit και θα περιοριστώ εδώ στη, στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έχουμε ασχοληθεί με τι επιπτώσει του Brexit στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά. Δεν ξέρετε ποιοι είναι, είναι οι κανόνε λειτουργία τη Επιτροπή μα. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε στο Συμβούλιο γι' αυτό. Έχετε την πρόθεση να είσαστε, να λάβετε δράση γέρος τώρα, ήδη, ακόμα και αν είναι νωρίς, ή θα περιμένετε το τι θα γίνει από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου για να αντιδράσετε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι ήδη. Ε, και το δεύτερο. Αυτό που αποσχολεί πολύ το κοινοβούλιο αυτόν τον καιρό είναι σαφώ το Brexit, αλλά υπάρχει άλλο ένα θέμα που είναι το κυνήγι των πουλιών στην ε, Μάλτα. Και γι' αυτό ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο για τους οικοτόπους των πτηνών. Και έχουν ήδη ακουστεί ανησυχίες για την ε, παρεκκλήσεις της Μάλτας από την Οδηγία για την Προστασία των Πουλιών, ιδίως για τα ορτίκια. Ε, εδώ Πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε αυτές τις ε, παρεκκλήσεις και τι θα κάνει η Μάλτα ώστε να διορθωθούν οι διάφορες ανεπάρκειες παρατηρούντας σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής και την εφαρμογή του. πρόκειται να ληφθούν μέτρα εν ώψη και τη ε, εαρινή ε, κυνηγετική περίοδου που πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα στη Μάλτα. Ευχαριστούμε κυρία Γκερλίν για τον φιλελευθέρος ο κ. Μαζουρόνης. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα καλή τύχη και για σας προσωπικά και για τη χώρα σας ε, στη διάρκεια του εξάμεινου της Προεδρίας σας. Έχω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη χρηματοδότηση της ανακαίνησης ε, των κτηρίων. Είμαι Λιθουανός. Μέχρι το 2012 η διαδικασία ανακαίνησης των κατοικιών ήταν κάτι που είχε παγώσει για δεκαετίες επειδή δεν υπήρχε επαρκής χρηματοδότηση. Δεν υπήρχαν αρκετά οικονομικά κίνητρα για να ε, υπάρξουν επενδύσεις σε πολυκατοικίες με διαμερίσματα. Το 2012 όμως η Λιωθανία ε, εισήγαγε ένα νέο οικονομικό μοντέλο και την αξιοποίηση και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έκτοτε λοιπόν πάνω από 2.000 πολυκατοικίες ε, ανακαινίστηκαν. Ωστόσο, ο αρμόδιος φορέας στη Λιθουανία ε, λαμβάνει περισσότερες αιτήσει από πολίτες για τον εξεχρονισμό και την ανακαίνιση. Δεν μπορεί να συγχρηματοδοτήσει όμως όλα αυτά τα αιτήματα. Θα είναι ε, προτεραιότητα στη Μαλτέζικη Προεδρία το πακέτο ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ε, στις κατοικίες. Οπότε θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποια μέσα, οικονομικά εργαλεία ή πρόσθετη χρηματοδότηση για να ενισχυθεί προσπάθεια ανακαίνησης των κτηρίων στις χώρες μέλη τη Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΕ, κυρία Κονέψινα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να δώσω συνέχεια σε αυτό που μόλις είπε ο συνάδελφος. Αναφέρατε τις προτεραιότητες σας, ε, μεταξύ άλλων ε, το, τη δεσμή μέτρων για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προβλέπετε το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων ε, του σημαντικού αυτού θέματος στο Συμβούλιο. Και επίσης, η Μάλτα θέλει να πετύχει την κοινή προσέγγιση πάνω στο θέμα αυτό. Η Σλοβακία δεν ε, πέτυχε συμφωνία για το σύστημα εμπορία εκπομπών και μου φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα είναι ακόμα πιο ε, επίμαχο. Πάντω, θα ήθελα πολύ να ενημερώσετε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, ε, όσον αφορά τον επιπερισμό της προσπάθειας και την μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Δεν κατάφερε η Σλοβακική Προεδρία να πετύχει γενική προσέγγιση πάνω στο θέμα αυτό και γι' αυτό σας ρωτώ. Πιστεύετε ότι θα έχετε εδώ την ε, δυνατότητα να σημειώσετε μεγαλύτερη επιτυχία και τι συγκεκριμένα σχέδια έχετε. Μπορούμε να υπολογίσουμε σε άνοιγμα του τριμερούς διαλόγου η Σλοβακική Προεδρία μας ε, είπε σχετικά με το Λούλου CF ε, και τον ε, επιμερισμό της προσπάθειας ότι θα πρέπει αυτά τα θέματα να εξεταστούν μαζί και ότι το νωρίτερο τον Μάρτιο θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο την θέση του Συμβουλίου. Πώς βλέπετε εσείς το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να έχετε επιτυχία ή πιστεύετε ότι όπως και η Σλοβακική Προεδρία δεν θα πετύχετε τίποτα. Εγώ προσωπικά θα απογοητευτώ εάν μπλοκαριστούν τόσο σημαντικά θέματα ακριβώς λόγω της θέσης του Συμβουλίου. Ο κύριος Αφρόντε από τους Πράσινους παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Ήθελα να αναφερθώ σε έναν από του στόχου που αναφέρατε, τον έκτο τη Προεδρία σα, για τι θάλασσε. Σχολιάσατε τη γαλάζια ανάπτυξη τη Σύνοδο 25 και 26 Απριλίου που θα ασχοληθεί με κάποια από τα θέματα αυτά της ναυτιλίας και της ναυσιπλοείας. Είστε από μια χώρα που προφανώς βασίζεται στη θάλασσα και μάλιστα τη Μεσόγειο. Και εγώ το ίδιο. Ε, οι ακτές μας είναι, ακτές της Μεσογείου. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι καταστροφική. Υπάρχουν θέματα που επικαλύπτονται η πρόσβαση στην αλία, το 90% των ευθυακών αποθεμάτων, οι συνέπειε των κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν πολύ σημαντικό τρόπο η χημική ρήπανση, η ρήπανση από στερεά υλικά όπως τα πλαστικά, οι επιθετικές δράσεις για την ε, εξερεύνηση του πυθμένα των θαλασσών για πετρέλαιο και άλλα ορυκτά, όλες αυτές είναι ενέργειες που ε, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη διακυβέρνηση λοιπόν εδώ, την οποία θα αναλύσουμε και θα εξετάσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, και με τον αρμόδιο επίτροπο, τον Επίτροπο Βέλλα, αλλά νομίζω ότι επειδή η Προεδρία σας ε, από ένα κράτος που ακριβώς είναι κράτος της Μεσογείου είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα. Και πολύ γρήγορα, επειδή δεν το σχολίασαν άλλοι ε, υπ' αυτή την έννοια, για τις κλιματικές αλλαγές, βεβαίως η συμφωνία ακόμα έφταστη γιατί μόλις ξεκινά και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διατηρήσει τον πρωτονιστικό της ρόλο. Όμως, Εάν δεν μου διαφεύγει, δεν αναφερθήκατε πέραν του ETS σε άλλες περιπτώσεις κατανομής των ε, αρμοδιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί για μείωση 40% στο 2030, αλλά δεν είναι ε, το μόνο πρόβλημα να μην ε, έχουμε αύξηση κατά δύο βαθμούς. Είναι πολύ περισσότερη προσπάθεια που χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να μου πείτε αν θα αναλάβετε επίγουσα δραστική, αν, θα κάνετε δραστικέ κινήσεις πριν το 2020 για του στόχου που είναι τόσο φιλόδοξοι και που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και τελευταίο ομιλητή για τον πρώτο γύρο. Η κυρία Δανανό από την ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μεταξύ των στόχων για το περιβάλλον, το πρόγραμμα της Μαλτέζικης Προεδρίας προβλέπει να προβλέψει μια αποτελεσματική οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα πόρου, αλλά και ανταγωνιστική οικονομία. Δύο ερωτήματα λοιπόν προκύπτουν. Πρώτον, δεν είναι επιτακτική ανάγκη η ανταγωνιστικότητα που ήδη αναφέρεται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν αποτελέσει ένα νέο κίνητρο αλλά που μπορεί να οδηγήσει τους παραγωγούς και τους βιομηχάνους μας να μετατοπιστούν σε ένα πλαίσιο πλήρους ανοίγματος της ε, οικονομίας μας και καμίας προστασίας από την Ευρώπη και έπειτα πώς μπορεί να συμφιλειωθεί απέτηση της ανταγωνιστικότητας με οικολογικούς στόχους που είναι όλο ένα και περισσότερο φιλόδοξοι ε, εν ώψη αυτής της ε, χωρίς ενδιασμούς διεθνούς του διεθνούς ανταγωνισμού που δεν έχει ενδιασμούς δεν είναι ένας αγώνας δρόμου αυτό χωρίς ε, ελπίδα και για την ε, χαμηλή κατανάλωση άνθρακα πόρους. Η Μαλτέζικη Προεδρία θα πρέπει να περιλάβει το σύστημα της ναυσιπλοείας ε, στο σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών. Δεν πιστεύετε ότι από αυτήν την έννοια θα πρέπει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή ε, Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον ILO που έχει, τον IMO που έχει την αρμοδιότητα για να δράσει τέτοια θέματα. Επίσης, το πρόγραμμα της Μαλτέζικης Προεδρίας δεν έχει λεπτομέρειες για το τι ε, κινήσεις θα γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, ποια είναι η θέση της Προεδρίας της Μάλτας για τη μείωση των εκπομπών ε, άνθρακα σε τομείς που δεν υπόκειται στο σύστημα ETS, λόγω χάρη τον κατασκευαστικό ή τη γεωργία. Και για τους στόχους μείωσης σε εθνικό επίπεδο, όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2016. Ποια είναι ακριβώς η θέση σας. Σας ευχαριστώ και τον προτέρων για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ. Προτείνω να απαντήσετε στις ερωτήσεις του πρώτου γύρου. Ο Υπουργό, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους ευρωβουλευτές για τις ευθείες και σημαντικές ερωτήσεις τους. Ε, κάλυψαν κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Φυσικά υπάρχουν επικαλύψεις. Θα προσπαθήσω όμως όσο γίνεται πιο σύντομα να διατρέξω τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Η πρώτη ερώτηση ήταν του Άιβο Μπέλετ. αναμενόμενο ήταν ε, να ακουστούν πολλές ερωτήσεις για το σύστημα επορίας εκπομπών. Το Κοινοβούλιο εκφράζει την αίσθηση του επίγοντος εδώ και το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις συζητήσεις με στόχο να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση όσο γίνεται ε, πιο σύντομα. Οι φιλοδοξίες είναι υψηλές και το Συμβούλιο Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις και να συνεχίσει να παίζει το ρόλο της ε, ως ε, σημαντικός και αξιόπιστος εταίρος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Συζητώνται όλοι οι τρόποι ενίσχυσης του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών. Έχουν υποβληθεί διάφορες ιδέες και προτάσεις. Με ρωτήσατε σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Συμβούλιο. Πολύ εύστοχη ερώτηση. Συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόοδο στο σημαντικό αυτό θέμα. Και επικεντρωνόμαστε στις βασικές εκκρεμότητες με στόχο να πετύχουμε γενική προσέγγιση όσο γίνεται πιο σύντομα. Υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες. Οι βασικότερες είναι οι εξής. Να έχουμε διατομεακό παράγοντα διόρθωσης, ενίσχυση ε, του συστήματος εμπορίας εκπομπών, ε, ε, αποτρέποντας και τον κίνδυνο με κατάσταση των εκπομπών του άνθρακα. όσον αφορά το θέμα της ναυτιλίας. Η Προεδρία βασίζεται στις εργασίες ε, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και εξετάζουμε και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει εδώ διεθνής διάσταση που ξεπερνάει τις ευρωπαϊκές προοπτικές διότι είναι θέμα διεθνούς εμπορίου και γι' αυτό είναι καλύτερο να συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς. Όπως άλλωστε προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ντάλια από τη Μάλτα έθεσε ερωτήσεις ε, σχετικά με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Η Συμφωνία του Παρισιού έχει τονίσει ιδιαίτερα τις δράσεις προσαρμογής ε, που νομίζω ότι δίνει νέα ορμή στην ε, συζήτηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε να υιοθετηθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2017. Δυστυχώς, ίσως ευτυχώς για μας, αλλά δυστυχώς θα πω παρόλα αυτά, μετά τη δική μας προεδρία. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε το σημαντικό θέμα της προσαρμογής ε, στην ε, αλλαγή του κλίματος ε, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το Άτυπο Συμβούλιο. Όπως είπα κατά την εισαγωγή μου, σκοπεύουμε να οργανώσουμε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών κατά το οποίο θα θίξουμε το θέμα αυτό. Άλλη σημαντική ερώτηση της συναδέλφου Μίρια Μταλή έχει να κάνει με το Euro 5 Η Μαλτέζικη Προεδρία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαπραγματευτεί πιθανές λύσεις για τα θέματα που εκκρεμούν ακόμα μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία όπως είναι η υποχρεωτική η εισαγωγή μετρητών ε, κατανάλωσης των καυσίμων. Αυτό και άλλα θέματα έχουν ήδη συμφωνηθεί επί Λουξεμβουργικής Προεδρίας. Επί της ουσίας φαίνεται να υπάρχει γενική συμφωνία. Με αυτήν την ε, ισχυρή βάση σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. Ε, πρέπει να ασχοληθούμε και με κάποια διαδικαστικά θέματα. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Το Brexit αναφέρθηκε από την κυρία Τζούλι Γκέρλινγκ. Περίμενα τέτοια ερώτηση κατά την ε, ομιλία μου, κατά την εισαγωγική μου ομιλία. Ανέφερα ότι περνάμε δύσκολες εποχές, ενδιαφέρουσες αλλά ιδιαίτερα δύσκολες και το Brexit είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν αναταράξεις. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να αναλύσουμε τις επιπτώσεις του Brexit. Πολλοί αναλύουν τις συνέπειες. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ βρετανό εκπρόσωπο, αλλά μόλις ενημερώθηκα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε ότι είναι απαραίτητο να γίνει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Στην Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων. για να ε, ε, επικαλεστεί το Ηνωμένο Βασίλειο το άρθρο 50. Αυτή λοιπόν ήταν η απόφαση και Φυσικά παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον το νέο αυτό θέμα που ανέκυψε. Η κυρία Γκέρλινγκ αναφέρθηκε και στις οδηγίες για την προστασία της φύσης. Στηρίζουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε να λάβουμε το νέο σχέδιο δράσης. Αφού υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωσή τη, ε, θα εξετάσουμε ποιο είναι ο πιο κατάλληλο τρόπο να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την Μάλτα. Συχνά μιλάμε εμείς οι Μαλτέζοι πολύ για τη Μάλτα, αλλά μου είπαν πριν έρθω εδώ εφόσον θα ομιλώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, ε, να μην επικεντρώνομαι ιδιαίτερα στην Μάλτα, αλλά βέβαια υπάρχει πάντα αυτή η τάση. Όσον αφορά λοιπόν το κυνήγι στη Μάλτα και άλλα τέτοια θέματα, ε, είναι θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε ε, κάποια άλλη στιγμή και προσωπικά διμερώς, δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μπω σε λεπτομέρειες. Θα σας πω ωστόσο ότι δεν θα επιτρέψω στην Μαλτέζικη νομοθεσία να προδικάσει τη θέση μου στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Επίσης, ε, ο κύριος Μαζουρόνης ε, έθεσε ερώτηση σχετικά με την ενέργεια. Η ενέργεια συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον ε, και γι' αυτό δεν τον κατηγορώ που έθιξε θέμα ενεργειακό στην συγκεκριμένη επιτροπή. Ωστόσο, το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο Συμβούλιο ε, Ενεργειακών Υποθέσεων. Και ο συνάδελφος μου, ο αρμόδιος υπουργός της Μάλτας, θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να απαντήσει εκείνο. Έχω σημειώσει την ερώτησή σα και θα τη μεταφέρω στον συναδελφό μου. Ο κύριος Μάρκο Αφρόντε από την πολιτική ομάδα των Πρασίνων. Είναι Ιταλός. Φόρεσα λοιπόν τα ακουστικά μου για να τον ακούσω, παρότι ε, μιλώ και εγώ Ιταλικά. Παρ' όλα αυτά θα απαντήσω στα αγγλικά. Μίλησε για ένα θέμα πολύ αγαπητό ε, στην Μάλτα που είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Προφανώς η Μάλτα είναι νησί, βρίσκεται στη μέση της Μεσογείου. Το θέμα της ε, θαλάσσης λοιπόν είναι τεράστιας σημασίας για τη Μάλτα. Όπω είπα, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων ε, της ε, Μαλτέζικη Προεδρίας, ε, τα ναυτιλιακά θέματα συμπεριλαμβανομένη της διαχείριση των ωκεανών, το έχουμε θέσει ως σημαντική προτεραιότητα στο θεματολόγιο μας. Κατά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος θα ασχοληθούμε με το κλίμα και με την ε, θαλάσσια βιοπικιλότητα και πόσο σημαντικό είναι να προωθήσουμε ε, την ε, υγεία, την υγεία ανάπτυξη των ωκεανών. Επίσης, φέτος το θέμα των θαλασσών ήταν σημαντικό και στο G7. Άλλωστε έχουμε και τον ε, στόχο βιώσιμη ανάπτυξης υπαριθμών 40 του θεματολογίου βιώσιμη ανάπτυξης. Ε, όλα αυτά λοιπόν ε, θα συζητηθούν κατά την διάσκεψη «Η ωκεανή μας» που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα. Στη Νέα Υόρκη είχα την χαρά να συμμετάσχω σε τέτοια υψηλή διάσκεψη. Και το καλοκαίρι του 2017 η πολύ σημαντική αυτή η διεθνής διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Βαλέτα, στη Μάλτα. Κατόπιν ε, είχαμε την κυρία Κατερίνα να Ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που προφέρω κάποια ε, επώνυμα. Και εσείς μάλλον θα βρίσκετε ακόμη πιο περίεργα τα δικά μας επώνυμα, τα μαλτέζικα. Δεν λέω ότι βρίσκω περίεργο το επώνυμό σας, απλά ε, δυσκολεύομαι να το προφέρω. Ελπίζω μέσα στους επόμενους μήνες ε, να βελτιωθεί η προφορά μου. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Η κυρία Κονέτσινα λοιπόν έθεσε ερώτηση παρόμοια με αυτήν της ε, κυρίας Ντάλη όπως ήδη ανέφερα, αναφερθότανε στο, στο CSR. Προφανώς το θέμα αυτό δεν είναι τόσο παλαιό όσο ε, το σύστημα εμπορία εκπομπών. Ε, ωστόσο, θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο πάνω στην πρόταση ESR με στόχο να πετύχουμε γενική προσέγγιση και σε αυτό το θέμα. Ποια είναι η κατάσταση εντό του Συμβουλίου. Συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα κράτη-μέλη για να προωθήσουμε τις συζητήσεις πάνω στα δύο βασικά θέματα. Ε, το σημείο εκίνηση ε, και τα μέσα ευελιξίας. Ε, όσον αφορά το θέμα Λουλουσιέφ, η Μαλτέζικη Προεδρία επίσης σκοπεύει να σημειώσει πρόοδο πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης παρακολουθούμε τη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άλλωστε είμαστε όλοι συνομοθέτες. Εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι δημοκρατική η διαδικασία και πολύ καλή η μέθοδος αυτή και γι' αυτό παρακολουθούμε από κοντά τα όσα συμβαίνουν εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατόπιν, ε, Ντοράνο, Όπω είπα, υπήρχε επικάλυψη μεταξύ κάποιων ερωτήσεων, ε, να μην επαναλαμβάνομαι. Νομίζω ότι απάντησα στι ερωτήσει σας. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Οι συνάδελφοι τώρα θα έχουν την ε, δυνατότητα πλήν των συντονιστών να που είναι και αυτοί τα δικά του. Ο κύριο Λίζε, Πρώτο. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την εισαγωγική του ομιλία. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω ένα ε, σημείο που ήδη αναφέρθηκε και κάτι που δεν αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά την εμπορία εκπομπών. Θα ήθελα να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο ε, είτε τώρα αυθορμήτως ε, ή όπως είπαν και οι συνάδελφοι τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ε, να λάβετε υπόψη σας αυτά που είπαμε η βιομηχανία ε, θέλει να υπάρχει ισχυρότερη προστασία κατά της διαρροής άνθρακα σε σχέση με αυτό που προτείνει η Κομισιόν και αυτό είναι προτεραιότητα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το ΕΛΚ είναι προτεραιότητα. Δεν θέλουμε μείωση ε, του επίπεδου φιλοδοξίας και έχουν γίνει διάφορες προτάσεις μεταξύ αυτών και αυτό που είπε ο κύριος Εβομπέλετ για την αεροπορία. να συμμετέχει στον επιμερισμό των βαρών ε, με μεγαλύτερο μερίδιο και αεροπορία. Σίγουρα η συμφωνία στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ δεν αρκεί με την πρόταση τη Κομισιόν υπάρχουν και άλλοι παράγοντε και άλλε παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και σας παρακαλώ να τα λάβετε αυτά σοβαρά υπόψη. Το δεύτερο είναι η αντοχή στα αντιβιωτικά ένα μείζον ζήτημα, αναφέρθηκε, είναι στον τομέα αρμοδιοτήτων Σα Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία σε ό,τι αφορά τη χρήση αντιβιωτικών στη γεωργία, να υπάρξει μια στρατηγική μείωση, δηλαδή όχι μόνο όπως έχει προτείνει η Κομισιόν να υπάρξουν κάποιε προτάσει από τα αντιβιωτικά, αλλά είναι πολύ σαφή η στόχη και να υπάρξει στρατηγική μείωση χρήση των αντιβιωτικών, ιδίω για τη Γεωργία, γιατί έχουμε το πρόβλημα ε, και τη διασύνδεση, τη στενή σχέση μεταξύ τη αντοχή ε, αντιβιωτικών ε, που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο και που χρησιμοποιούνται για τα ζώα. Και θα πρέπει. <clears throat> Και θα πρέπει να λάβετε υπόψη, πιστεύω, αυτό το θέμα στι διαπραγματεύσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου και να προωθήσετε θετικά τα πράγματα. Ξέχασα να πω στους συναδέλφους, λέει η Πρόεδρος, ότι ένα λεπτό είναι πλέον ο χρόνος ομιλίας, ώστε ο Υπουργός να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Η κυρία Μποναφέ είναι επόμενη. Ευχαριστώ Πρόεδρε Υπουργέ, καλή ε, τύχη και συγχαρητήρια για το φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει υποβάλει η Μαλτέζικη Προεδρία γενικότερα για τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη και όλος ιδιαίτερος και για τα τόσο πολλά ζητήματα που απασχολούν τη δική μας Επιτροπή. Ήδη απαριθμίσατε διεξοδικά τις προτεραιότητές σας. Εγώ λοιπόν δεν έχω παρά να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την προτεραιότητα που θα δώσετε στην κυκλική οικονομία και στο σχετικό ντοσχέ. Σωστά τα είπατε. Από τη μια πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντο, από την άλλη όμω ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να ε, αναθερμάνουμε και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Σωστά το είπατε. Ψηφίσαμε πρώτη φορά για τον ντοσχέ αυτό στην Επιτροπή μα. Είδατε ότι εγκρίθηκε με ευρεία και ξεκάθαρη πλειοψηφία θα έλεγα. Και ε, η θέση μα είναι φιλόδοξη αλλά και πραγματιστική. Δηλαδή, Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε για μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση επί του θέματος και προς αυτό το σκοπό πρέπει να πω ότι η γενική, ε, το γενικό κλίμα που έχουμε στις συνεργασίες μας με τη Μαλτέζικη Πρόεδρε είναι πολύ θετικό. Σε μερικά ζητήματα μόνο υπάρχουν αποκλήσεις, κυρίως στους στόχους και τη μέθοδο υπολογισμού, αλλά δεν ε, μας διαφεύγει ούτε εμένα ούτε από εσάς το ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε αυτό το ντοσχέ. Η αξιοπιστία της Ευρώπης έχει να κάνει με το τι πορεία θα πάρει το όλο θέμα. Εάν μπορέσουμε να προβλέψουμε ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο, δίνουμε στους επενδυτές την ευκαιρία να το κάνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και από τη δική μου πλευρά θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μία μάλλον και οι δύο αφορούν την αυτιλία, το θαλάσσιο τομέα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Διεθνή Αυτιλιακό Οργανισμό που αναφέρατε. Αναφερθήκατε επίσης και στη ΔΟΠΑ και, τις, ε, ε, και το ETS. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμό δεν ε, συμμετείχε ούτε σε εργασίες της των Παρισίων στο πλαίσιο της ΚΟΠΕ και αυτό ήταν ένα λάθος. Ε, γιατί θεωρώ ότι και τα πλοία ε, πρέπει να λαφθούν υπόψη, θα πρέπει να υπάρξουν ε, κατευθείαν γραμμές για τιμή των εκπομπών και από τα πλοία. Εσείς πόσο θα μπορούσατε να προωθήσετε αυτό το αίτημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για την Βαλτική, για παράδειγμα, 0,1 εκπομπές μόνο και για τη Μεσόγειο καλό θα ήταν και για τον αέρα εκεί γενικώ να βελτιωθεί η κατάσταση. Το δεύτερο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα έχει να κάνει με την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών Ocean Governance. Είπαν οι κάποια πράγματα. Η Μάλτα είναι ε, θαλάσσιο κράτος. Είστε σε επαφή με τη ΣΥΠΑ, ο Ντόναλτ Κραμπ είπε για τους στόχους της COP21 ότι θα επαναχωρήσει και δεν θέλει και τόσο πολύ να ασχοληθεί με το ε, κλίμα. Πόση επιρροή θα μπορούσατε να ασκήσετε στο πλαίσιο της Προεδρίας που έχετε, να επηρεάσετε λίγο τις ΥΠΑ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now, Mr. Linz. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κατά την εισαγωγή σας ε, αναφερθήκατε στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και αναφερθήκατε επίσης στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, καθώς και στον κανονισμό LULUCF. Είπατε ότι θέλετε να πετύχετε πρόοδο πάνω στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας σας. Θα με ενδιαφέρε να μάθω πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Μέχρι μέσα Φεβρουαρίου πρέπει να υποβάλω την ε, έκθεσή μου εδώ. Έχω την εντύπωση ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν πολύ θέσεις. θέσει. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τα νότια κράτη-μέλη, ποια θέματα βρίσκουν εδώ ιδιαίτερα σημαντικά. Και τελευταία ερώτηση, πώς βλέπετε την ευελιξία των 280.000 τόνων. Ευχαριστώ. Thank you, thank you, Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τους φιλόδοξους στόχους σας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους ε, στόχους ε, της αναβιώσιμης ανάπτυξης, που είναι για μας μια πρώτη προτεραιότητα. Τρεις ερωτήσεις για το φινικέλαιο. Πολύ πρόσφατα είδαμε ότι υπήρξε διόγκωση της μη διώσιμης παραγωγής φινικελαίου Κάτι που έχει επίπτωση και στο κλίμα. Η έκθεση Globium από την οργάνωση αυτή δείχνει πόσο σοβαρός είναι αυτός ο αντίκτυπος. Τι μέτρα θα λάβει λοιπόν η Προεδρία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να υπάρξουν αντικίνητρα για την παραγωγή μη βιώσιμου φινικελαίου και επίσης για την κατάσταση διεθνώς. Ο πρόεδρος Τραμπ θα κοιτάξει στα θέματα της, ε, των κλιματικών αλλαγών να, ε, θα αφήσει σίγουρα καινή την πρωταγωνιστική θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τι θα κάνει για την πραγματική ανάγκη να διτηρηθεί ο ρυθμός της προόδου αμύωτος για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστούμε ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που βρήκατε χρόνο να έρθετε εδώ. Ευχόμαστε και από πλευρά της NGL ε κάθε επιτυχία στην ε, Μαλτέζικη Προεδρία για το επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με τον κανονισμό για τα πτηνά, καθώς και για το κυνήγι ε, πτηνών στη Μάλτα. Αλλά η συνάδελφος ήδη έθεσε το θέμα αυτό, γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Προφανώς ε, γνωρίζετε ότι η μαζική κτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά στην ε, ε, αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη λόγω των εκπομπών. Αυτές οι εκπομπές από τον γεωργικό τομέα δεν μπορούν να αγνοηθούν πια. Η γεωργική πολιτική όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπει αύξηση της παραγωγής, ε, ενώ θα ήταν πιο λογικό να στοχεύσουμε στην μείωση της παραγωγής. Αυτό το θέμα συνδέεται άλλωστε και με τα ανθεκτικά μικρόβια. Η Μαλτέζικη Προεδρία έχει σκοπό να ε, θίξει αυτό το μη δημοφιλές θέματα. Έχετε την τόλμη ε, να, ε, να εισηγηθείτε αλλαγές στον τομέα της γεωργικής πολιτικής ή θα συνεχιστούν τα πράγματα όπως μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πύρη. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο Όσον αφορά το επόμενο εξάμεινο, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτά που είπε ο κύριος Υπουργό, αλλά υπάρχει ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για τις κάτω χώρες. Ε, έχουμε το θέμα των ε, νητρικών αλάτων. Ε, δεν ξέρω αν ακούει ο Υπουργό, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα που θέλω να θίξω. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Το θέμα που θέλω να θίξω είναι πολύ σημαντικό στις κάτω χώρες. Έχει να κάνει με την οδηγία για τα νητρικά. Οι κάτω χώρες έχουν ε, κλίμα διαφορετικό από τη Σικελία ή τη Μάλτα. Και έχουμε πρόβλημα λόγω των ε, παρεκκλήσεων που προβλέπονται. Η Μαλτέζικη Προεδρία μήπως ε, θα μπορούσε να προβλέψει συζήτηση σχετικά με την παρέκκληση για το 2017. Μπορείτε να μας στηρίξετε και συγκεκριμένη ερώτηση. Μπορείτε να μας απαντήσετε πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Χιλιάδες αγρότες ε, δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκριλάκ. E, e, e, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Χαίρομαι που σε αυτή την απαρίθμηση ε, αναφέρεται και την κυκλική οικονομία. Έχω δύο ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένε. Διότι μεταξύ άλλων η Μάλτα είναι μεταξύ αυτών των κατομελών που έχουν προβλήματα. Προβλήματα με τα χήτα. Την αποκομιδή των ε, αποβλήτων και είναι και μια μεσογειακή χώρα που πρέπει να ασχοληθεί και με τα θέματα των θαλασσίων αποβλήτων, των αποβλήτων στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν που θέλω να μου πείτε είναι πόσο έχει ενδιαφερθεί η Μάλτα για να στηρίξει την πρότασή μας για να μειώσουμε την κατασπατάληση τροφίμων κατά 50% στο 2050. Και επίσης αυτό συμβαδίζει με όσα είπε η Μαλτέζικη Προεδρία και η εκπρόσωπή της για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης για την ψηφοφορία που είχαμε σήμερα το πρωί ε, και όταν μιλάμε για την ε, διαλογή των ε, αποβλήτων, τον ιεράρχησή τους, δεν είναι ξεκάθαρο ποια μέθοδο θα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό ήθελα την γνώμη του Υπουργού σχετικά και το κατά πόσον αυτό θα αποτελέσει μέρο των προτεραιοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας. Θα στηρίξει τη δουλειά μας εδώ στο Κοινοβούλιο η Μάλτα, διότι το πρόγραμμα είναι ούτως ή άλλως πολύ φιλόδοξο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φλόρεντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προεδρεύοντα. Καλώς ήρθατε. Προσωπικά Ε, υπάρχει κάτι που μας συνδέει στο 55ο σε προεδρεύον του Συμβουλίου με τον οποίο έρχομαι σε επαφή και πρέπει να σας πω ότι έχω ακούσει όλο αυτό το διάστημα πολλές διαφορετικές ομιλίες. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι σχεδιάζετε για το επόμενο εξάμεινο και θα σας στηρίξουμε σίγουρα. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο είναι αυτό που θα μπορούσατε να συνεισφέρετε ιδίως ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής γιατί υπάρχουν πολλά που έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Έχουν αποφασίσει την κυκλική οικονομία σήμερα. Πολύ σημαντική απόφαση. Όμως ε, η οδηγία 20 χρόνια ε, εργάζομαι πάνω σε αυτό το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί με λογική. Αυτό θα πρέπει να το επεξεργαστούμε. Τι προβλέπετε λοιπόν για τα κράτη-μέλη όπως είναι η Γερμανία, και πολλοί άλλοι σε πολύ ωραίες ε, γειτονικέ χώρες ε, που δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά και Ρουμανία και Βουλγαρία σε σχέση με την πολιτική γειτονία. Θα πρέπει να δείξετε σθένος ε, και θα πρέπει να πιέσετε την Κομισιόν ώστε τελικά να κάνει αυτό το οποίο έχουν αποφασίσει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Γνωρίζω ότι δεν είστε στην Κομισιόν. Όμως θα ήθελα να σας παροτρύνω για κάτι. Έχω δει και χώρε μεγάλες χώρες που έχουν κάνει πολλές υποσχέσει και δεν έχουν κάνει τίποτα στην πράξη. Έχω δει όμω πολύ μικρές χώρε να έχουν, κινήσει, να έχουν βουνά. Επομένως, ε, καλό είναι ε, κάθε φορά να πιέζετε και να λέτε στην Κομισιόν τι πρέπει να εφαρμόζει. Εγώ είμαι Γεωργός. Ε, άκουσα την κυρία Σράιερ Πύρικα και υπήρξε, κάποιες αντιρρήσεις για αυτά αλλά έχουμε ένα νόμο το 1981 και καταγγέλει τη Γερμανία. Αν αύριο ε, τρέξω ε, πιο γρήγορα, ε, πληρώνω πρόστιμο την επόμενη μέρα Είπα στο το δικαστήριο. Δεν μπορούμε να αργούμε τόσο πολύ. Ελπίζω να έχετε κίνητρα και να προχωρήσετε αυτά τα θέματα. Thank you very much, Mr. Florence. Um, next speaker, Mr. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και να συμφωνήσω με αυτά που είπε νωρίτερα ο Νόρμπερτ Λίνς σχετικά με τη σημασία του Λούλου CF της ε, χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και Σε Πρόταση που ε, έλαβε το Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Λίνς είναι εισηγητής και εγώ είμαι σκιώδη εισηγητής για ε, την ομάδα των σοσιαλιστών. Και έχει αναφερθεί ότι μπορεί να ψηφοδρομήσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά ε, την ε, αντιμετώπιση τη αλλαγή του κλίματο, που μπορεί να σημαίνει ότι το υπόλοιπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να κάνει περισσότερα και γι' αυτό το θέμα τη Λουλουσιεφ θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό. Η Μάλτα βρίσκεται στον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το μικρότερο ποσοστό κάλυψης από τάση ε, στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι επίκριση, είναι γεγονός. Ε, παρακαλώ όμω να μην ξεχάσετε τον ρόλο και τη σημασία της δασοκομείας ε, στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Ε, θα το δείτε αυτό και στην πρόταση LULUCF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ελπίζουμε να βελτιώσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και το θέμα δεν είναι μόνο η δασοκομεία, είναι και η παραγωγή ξυλίας, ε, η αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Ό,τι μπορέσετε λοιπόν να κάνετε στο τομέα της δασοκομείας ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για να προωθήσετε τη χρήση ξυλίας ε, και την ε, φύτευση περισσότερων δέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματα που μπορούμε να επικροτήσουμε. Η κυρία Αγιούσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πολύ σύντομα θα αναφερθώ στην οδηγία έχουμε κάποιες προτάσεις κομισιών για παράτηση παζινίας το 2020, ό,τι αφορά τα έτη 2017-2018 τώρα. Οι εκπομπές είναι πιο χαμηλές. Αυτό οφείλεται στην κρίση βέβαια όμως. Τα κράτη-μέλη χάνουν κάποιες εκπομπές για τις οποίες είχαν δικαίωμα και πιστεύω ότι το 2020 θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε δηλαδή να αυξήσουμε το στόχο πέραν του 30% αλλά να το δούμε τότε η αντιστάθμιση τώρα στο μηχανισμό ευελιξία για τη χρήση των γιών και των δασών. Είναι ασυμμετρική. Αν αυξάνονται οι εκπομπέ θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Όμως αυτή τη στάθμιση και ο υπολογισμό περιορίζει τα 280 εκατομμύρια τόνους ε, διοξιδίου του άνθρακα, αλλά μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο το τμήμα που χρησιμεύει για την αντιστάθμιση πλονάσματο. Επομένω, ο μηχανισμό ευελιξία είναι μόνο στο χαρτί ουσιαστικά και δεν αξιοποιείται στην πράξη επαρκώς. Γι' αυτό αν έχετε κάτι να πείτε, ευχαριστώ. Thank you very much. Colleagues now, Minister, a lot of questions. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, συναδέλφους. Κύριε Υπουργέ, μακρύς ο κατάλογος των θεμάτων. Παρακαλώ, όποτε είστε έτοιμος. Ναι, θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Σε κάποια θέματα ίσως να είμαι λίγο πιο αόριστος από ό,τι σε κάποια άλλα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Σε ό,τι αφορά τον Ντόναλτ Τραμπ, για παράδειγμα, και τους ορισμούς και τα λοιπά, δεν υπάρχει αφιβολία ότι θα υπάρξει απόσταση από τη Συμφωνία των Παρισιών. Είπα, ήταν σημαντικό ε, εταίρο. Ε, είχε συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της Συμφωνίας των Παρισίων και την αλλαξή σχέση της ε, συνθήκης. Έχουμε και την αναγγελία ένα χρόνο πριν από την COP21, είπα και Κίνας, δύο πολύ σημαντικών εκπομπών των ε, χωρών που εκπέμπουν πολύ σημαντικές ε, εκπομπές και γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε ακόμη να προδικάσουμε τις αλλαγές στο πώς θα συμμετέχει στα διεθνή δρόμενα πλέον ε, η Αμερική, όμως σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούμε υπό διαφορετικά γεωπολιτικά σενάρια αυτά μπορούσαν λοιπόν να αλλάξουν δραματικά γεωπολιτικέ συνθήκες, πράγματι. Δεν είναι πολύ ακόμη ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να οργανωθεί επ' αυτού. Υπήρχε μια σημαντική ερώτηση από τον κύριο Ντάβορ Σκρέλακ για το νομοθετικό πακέτο για τα απόβλητα. Είναι ένα θέμα που φαίνεται όμως να προχωρά και αρκετά ομαλά σε ό,τι το επίπεδο φιλοδοξία. Ω Συμβούλιο, ω Προεδρία συγκεκριμένα, στάζουμε ορισμένε επιλογέ ώστε να έχουμε μια ρεαλιστική αλλά και φιλόδοξη προσέγγιση για όλα αυτά τα θέματα. Οι επιλογέ αυτέ συζητούνται και στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Αλλά βέβαια προ το πάνω στα χέρια των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα διατροφικά τα κτλ. Και φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την ε, άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Κάποιο σχόλιο, ο Πέτερ Λίζε τώρα, με κάποιες πτυχές, αρκετά τεχνικές θα έλεγα, Και καλά έκανε ο κύριος Λίζη γιατί πρέπει να δούμε την πρόταση ε, και τα στοιχειώδη αυτά θέματα θα τα μελετήσω. Είναι κρίσιμα ζητήματα και θα τα μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και με περισσότερη λεπτομέρεια. Σε ό,τι αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τα αντιβιωτικά θέλουμε ο κανονισμός ε, να παραμείνει φιλόδοξος και η σχετική ρύθμιση. Σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων, ε, στρατηγική μείωση ε, της χρήσης των αντιβιωτικών. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τη χρήση για τη μικροβιακών φαρμάκων. Και θα δούμε στα πλαίσια αυτού του κανονισμού και της τροπολογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τεχνικής πλευράς με στόχο να έχουμε μια διαπραγματευτική εντολή για το θέμα αυτό στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Κυρία Μποναφέ, για το μυθικό πακέτο για τα απόβλητα, φαίνεται ότι οδηγείται σε αίσιο πέρα στο θέμα, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την τελική ψηφοφορία. Θα λάβουμε υπόψη την θέση του Κοινοβουλίου. Επί του θέματος σίγουρα θα συνεργαστούμε. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο σε επίπεδο Συμβουλίου, εργαζόμαστε με όλα τα κράτη-μέλη για να προωθήσουμε τα βασικά ζητήματα, όπως είναι οι βασικοί ορισμοί, οι στόχοι και ο υπολογισμό. και οι σχετικοί κανόνες. Σε ό,τι αφορά το ΛΖΕΦ πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά. Γιατί πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας. Το Συμβούλιο θα διαφερθεί μεταξύ άλλων ιδιαίτερα και για τα επίπεδα αναφορά, ό,τι αφορά τα δάση. Αυτό είναι η απαραίτητα αφετηρία, πιστεύω, για το μελλοντικό μας έργο σε αυτό το τομέα. σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ευελιξία. Δεν έχουμε καταλήξει στο Συμβούλιο ακόμη σε ό,τι αφορά το Λουλουσιεύ για τα 280 εκατομμύρια τόνους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο όλων των ευελιξιών που προβλέπονται στον τομέα αυτό. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει έμφαση σε αυτές τις ε, πιστώσεις, σε αυτά τα δικαιώματα. Ο κύριος Μπρένεν, θέλω να τον ευχαριστήσω, έδειξε τον ενδιαφέρον και ο ίδιος για αυτό το θέμα. κυρία Πύρικ ε, βέβαια έκανε μια δική αναφορά στην Ολλανδία. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες και τις ενστάσεις. Το Συμβούλιο θα αναλύσει οποιασδήποτε αναφορές εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις που θα του υποβληθούν. Δεν έχουμε όμως ακόμη επιτάπητος μια σχετική ε, τροποποίηση οδηγίας για τα... Θα, θα δούμε. Φαντάζομαι το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί ούτως ή άλλως σε επίπεδο συμβουλίου. Για την κτηνοτροφία, ε, την εντατική την ε, εκτροφή, την εκτροφή ζώνη ήταν ένα θέμα και αυτό που προέκυψε, έχει να κάνει και με την αλλαγή του κλίματος. Βέβαια, χρήση των γεών. Μπορεί να θεωρηθεί και κτηνοτροφία χρήση γης σε έναν βαθμό. Και θα το δούμε και από την προοπτική του Λουλουσίεφ. I would, um, Για να ολοκληρώσω. Σημειώνω αυτό που είπατε ότι πολλέ φορέ πολλά λέγονται και σε επίπεδο συμβουλίου και σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλά δεν υλοποιούνται. Αυτό είναι ένα θέμα, πράγματι. Οι δομέ του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δημοκρατικέ Σε επίπεδο Συμβουλίου υπάρχει διαμεσολάβηση τη Προεδρία κάθε φορά που προσπαθεί να διαπραγματευτεί συμφωνίε. Επίση υπάρχουν διαφορετικέ ομάδε, διαφορετικέ ιδέε και προτεραιότητε σε επίπεδο ε, κοινοβουλίου. Άρα η δημοκρατική διαδικασία είναι ακόμα πιο δύσκολη εδώ από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Διότι απαρτίζεται το κοινοβούλιο από 28 ανεξάρτητα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό είναι το τίμημα τη δημοκρατία. Ο Γούσταν σημαντικότατο πρωθυπουργό, είπε κάποια στιγμή ότι η δημοκρατία μπορεί να μην είναι η ιδεώδης μορφή διακυβέρνησης, αλλά η δημοκρατία και η υπομονή, η διπλωματία συγγνώμη, και η υπομονή είναι αρετές για να ε, έχει τα καλά αποτελέσματα αυτή, αυτός ο θεσμός. Σας ευχαριστώ για τα επικοδομητικά ερωτήματα και θα συνεργαστώ με πολύ μεγάλη χαρά τους επόμενους μήνες μαζί σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Minister, and I wish... Ευχαριστούμε Υπουργέ. Καλή τύχη στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Ελπίζουμε στην αρμονική συνεργασία μας και ελπίζουμε και εμείς στη στήριξή σας. Α, χειροκροτήσουμε τον Υπουργό. Έτσι μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη της πρωινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε το απόγευμα στις 3.